Τα πρακτικά της συνεδρίας 16ης Φεβρουαρίου της διάθεσή σας υπάρχουν αντιρρήσεις. Όχι. Οπότε εγκρίνονται τα πρακτικά. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ε, στην συνεδρίαση της ε, της 1 Μαρτίου 2012 παρέλαβε τις νέες εντολές των βουλευτών. Πρόκειται για τον Νίκο Χρυσόγελο από τις 2 Φεβρουαρίου, του Φιλ Μπάνιαν από τις 6 Φεβρουαρίου και της κυρίας Έμα Κοστέλο από τις 15 Φεβρουαρίου. Προτείνω να εγκρίνουμε αυτές τις εντολές. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι, οπότε εγκρίνουμε την κυριότητα αυτών των εντολών. Ο κύριος Ρότζερ Χέλμερ μου είπε πως δεν